κρατήσετε κάποια ησυχία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρούμε πάρα πολύ θετική την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να ε, επιληθεί αυτό το πρόβλημα που είναι κατεπήγον όσον αφορά το να μην μεντάνει τον πρόεδρο του Σουδανικού Παρατηρητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως θυμάστε, συνελήφθη από τις διοικητικές αρχές της ε, ασφαλείας το Δεκέμβριο του 2014 και από τότε βρίσκεται σε απομόνωση στα πλαίσια της εκστρατείας της ε, κυβέρνησης κατά του αποκαλωμένου Σούνταν Κόλ. Ήταν δημοκράτης και επίσης εκπροσωπούσε κάποιες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών του Κεμβρίου. Οπότε ήταν μέλος της αντιπολίτευσης που είχαν ε, σηκωθεί τη κυβέρνηση. Για μένα είναι ένα ε, πρόσωπο πάρα πολύ ειδικού ηθικού βάρου. Ήταν ε, συνήγορο για πάρα πολλού από την ισχυρή των πολιτών, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έδρασε και στα δικαιώματα του. Το 2013 είχαμε μια, του, του απονείμαμε ένα βραβείο για τις δραστηριότητε του. Οπότε και απαιτούμε από την Σουδανική κυβέρνηση άμεσα να τον απελευθερώσει και αυτόν και τους άλλους πολιτικούς κρατουμένους. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας στο Χαρτούμ έχει επαφή με την οικογένειά του και συζητά ε, και βρίσκεται σε μια σειρά επαφών για τον Μεντάνη γιατί αυτό δεν είναι καμία παραβίαση μόνο του συντάγματος και του δικαίου στο Σουδάν, αλλά επίση αποτελεί καταπάντηση τη ελευθερία έκφραση, κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με τι διεθνεί αρχέ διαλόγου του ε, διεθνούς δικαίου, κάτι το οποίο είχε ασπαστεί στην αρχή της χρονιάς η κυβέρνηση του Σουδάν, οπότε θα πρέπει να μην έχουμε ε, ένα τέτοιο κλίμα καταπίεσης και καταστολής για τους πολίτες και θα πρέπει να είπαν να καταθέσουν τα όπλα και επίσης ε, από τις 20 Οκτωβρίου προκύπτουν τα συμπεράσματα σε σχέση με την κατάσταση των δικαιωμάτων στο Σουδάν που μας ανησυχούν πάρα πολύ. Η κατάσταση είναι ε, πάρα πολύ αυταρχική, καταστολές, σύλληψη, συλλήψεις ε, δημοσιογράφων, αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε τέτοιο είναι το πολιτικό κλίμα, έχουμε πάρα πολλές ελέγχους, έχουμε ε, λογοκρισία στον Ταρφούρ, στον ε, Ραζιονίλο και οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε επίσης αδιάκριτες ε, ε διενέργειες βομβαρδισμών κατά μάχων, οπότε χρειάζεται τώρα να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί όλα αυτά γίνονται σε ατιμορρησία, οπότε θεωρούμε πάρα πολύ σχετική αυτή την κατάσταση και επομένως θα πρέπει να δούμε το ότι η Αφρικανική Ένωση και ο πρόεδρος Μπεκί είχε αναλάβει κάποιες προσπάθειες για διάλογο την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς καμία επιτυχία. Σας διαβεβαιώ ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και η ειρήνη θα συνεχίσουν να αποτελούν δική μας προτεραιότητα και θα είμαστε επομένως συνέχεια σε επαφή με τις εμπλεκόμενες Σουδανικές Αρχές. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και με την ευκαιρία από πλευρά της ε, ε, Ιταλικής Προεδρίας θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά και καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντελαβέντοβα και εμείς από πλευρά μας σας ε, ευχαριστούμε για την προσπαθειά σας και αντευχόμαστε πέρα τη ζητήσεις.